Yes, of course. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε λοιπόν το δεύτερο αυτό τμήμα των, της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής. Δεύτερο μέρος σήμερα το πρωί. Μέχρι τις 11.30. Ε, στις 11.30 θα έχουμε την συνάντηση των συντονιστών. Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη για σήμερα σήμερα το πρωί που εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο της συνεδρίασής μας είναι η συνάντηση τον κύριο Ήταλα επικεφαλής δηλαδή του ελεγκτικού συναδρίου και για τις διοργανικές σχέσεις σε σχέση ακριβώς με το ελεγκτικό συνέδριο και εμάς. Ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μας και επιτρέψτε μου να επαναλάβω, να υπενθυμίσω ότι θα επικαιροποιήσει, θα ενημερώσει τα μέλη για τη συνεργασία μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και πώς μπορεί να ενδυναμωθεί το εγχείρημα της εξέτασης και του ελέγχου από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως γνωρίζετε θέλουμε να καταλήξουμε σε καλύτερο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό καμιά φορά σημαίνει ότι φυσικά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τον έλεγχο στο σκέλος του ελέγχου. Η ε, έκθεση για παράδειγμα ελέγχου εφαρμογής θα είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και ο κ. Σίταρα θα συζητήσει επίσης το πρόγραμμα εργασιών για το 2015 του Ελεκτικού Συνεδρίου, ιδιαίτερα και την έκτακτη ειδική έκθεση που ε, προετοιμάζει το ελεγκτικό συνέδριο. Να σας υπενθυμίσω ότι οι έκτακτες ειδικέ αυτές εκθέσεις αφορούν τα αποτελέσματα επιλεκτικών ελέγχων δειγματοληπτικά σε συγκεκριμένα θέματα. Δύο από αυτά τα σκέλη. Έλεγχος της, το θέμα των ενέργειας και ενεργειακών εφοδιασμού. και όσον αφορά και την πυρηνική ασφάλεια, θέματα πυρηνικής ασφάλειας και το θέμα φυσικά της αποτελεσματικότητας της χρήσης των κονδυλίων, των κοινοτικών κονδυλίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον πιο σωστό τρόπο και να ελέγχονται και να εξετάζονται οι διάφορες χρήσεις. Χρησιμοποιώντας αυτά τα κονδύλια και δαπανώντας τα πώς θα δαπανούμε και τι κάνουμε, ιδιαίτερα και για την έκθεση εφαρμογής και υλοποίησης. Η σημερινή λοιπόν ανταλλαγή απόψεων θα βοηθήσει να μπορέσουμε να κατανοήσουμε από πλευράς του ελεγκτικού συνεδρίου τι συμβαίνει και να μπορέσει έτσι να φτάσει η αποτελεσματικότητα αυτή μέσω αυτών των δράσεων, μέσω του προγράμματος εργασίας των ελεγκτών του ελεγκτικού συνεδρίου σε αποτελέσματα. Σας δίνουμε λοιπόν, ε, υπάρχουν προτάσεις λοιπόν που θα διατυπωθούν και στην αρχή αν μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε μια εισαγωγή και να κάνετε τα πρώτα σας σχόλια έχετε τον λόγο κύριε Ιταλά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ήτρε. Με ιδιαίτερη ευκαιρία προσφωνώ τα μέλη αυτής της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και θα ήθελα μια σύντομη εισαγωγή να δώσω και μετά θα ακούσω τις προτάσεις και ιδέες σας και αν υπάρχουν ερωτήσεις θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Το πρώτο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι είναι ένα ανεξάρτητο σώμα ελεγκτών το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν είμαστε τμήμα ή σκέλος των εσωτερικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε είμαστε σκέλος ή τμήμα κάποιου άλλου θεσμικού οργάνου. Πρέπει λοιπόν από πλευράς εντολής μας ασκώντας τις εξουσίες ελέγχου και εφαρμόζοντας σε σχέση με τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού προϋπολογισμού να ενημερώνουμε και το Ευρωκοινοβούλιο. Όσο καλύτεροι είμαστε σε αυτό το έργο, τόσο καλύτερα διασφαλίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο από τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητές μας στοχεύουν στο να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση. Να επικεντρωθούμε στα τελικά δηλαδή προϊόντα βελτίωσης ε, των λογιστικών στοιχείων και του τμήματος εκείνου που αφορά την αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, να μπορέσουμε να συντονιστούμε με τους εταίρους μας, ώστε να μεγιστοποιηθεί η λογοδοσία και ο έλεγχος πιο συγκεκριμένα Είμαστε δεσμευμένοι για να ε, παράσχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα μέσω των δράσεών μας που θα βοηθήσουν το Κοινοβούλιο. Να βοηθηθεί δηλαδή η χρήση ε, των κονδυλίων, η χρησιμοποίηση των κονδυλίων. Αλλά όλα αυτά δεν επαρκούν αν δεν τα χρησιμοποιούν οι αρμόδιοι για την πολιτική. Η δική μας προσπάθεια για την βελτίωση της λογοδοσίας και υπευθυνότητας εξαρτάται από τους άλλους εταίρους μας, παράδειγμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να βελτιωθεί αυτή η συνεργασία με τους κυριότερους εμπλεκόμενους, ξεκινήσαμε με το Ευρωκοινοβούλιο εξετάζοντας τις δυνατότητες βελτίωσης των δράσεών μας. Και ποια είναι τα προϊόντα μας, τα λογιστικά και ελεγκτικά. Η ετήσια έκθεση είναι το πιο σημαντικό που κάθε χρόνο αρχές Νοεμβρίου δημοσιεύεται. Επίσης ελέγχουμε τους λογαριασμούς 50 οργανισμών και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων φορέων. Έτσι λοιπόν πάνω από το ίμιση των δικών μας πόρων αναλώνεται σε αυτές τις δράσεις. Θα ήθελα όμως περισσότερο να μιλήσω σήμερα για τις δραστηριότητες που το όνομα δεν λέει και τόσα πολλά σχετικά προτάθηκε να αλλάξουμε τον τίτλο, το όνομα, ώστε να αντανακλώνται αυτές οι δραστηριότητες, εκθέσεις επιδόσεων, performance reports, για την αποτελεσματικότητα, την εξοικονόμηση, τον πιο σωστό τρόπο εφαρμογών ευρωπαϊκών κοινοτικών πολιτικών και προγραμμάτων. Value for money reports αποκαλούνται συχνά, δηλαδή αξιόλογες εκθέσεις που αξίζουν τα χρήματά τους. Σε αυτό θα δώσουμε περισσότερους πόρους εφεξής. Η δεύτερη μακρότερη πρόθεσμη, μακροπρόθεσμη προτεραιότητά μας είναι η συνεργασία και έχουμε δύο φυσικά επίπεδα διεξαγωγής αυτής της συνεργασίας. Πρώτον, όταν σχεδιάζει τις προτεραιότητες ελέγχου το, το ελεγκτικό συνέδριο για το επόμενο έτος και δεύτερον όταν δημοσιεύονται οι εκθέσεις ελέγχου. Εφέτος ξεκινήσαμε μια νέα διαδικασία. Ο πρόεδρος του ελεκτικού συνεδρίου συμμετέχει σε συνεδριάσεις ώστε να υπάρχει διάλογος με τους προέδρους των κοινοβουλευτικών επιτροπών του Κοινοβουλίου ώστε να κατανοήσει το έργο των κυριότερων πεδίων πολιτικής. Κατά τη διάρκεια και μετά αυτή τη συνεδρίαση που είναι σε 9 Ιουνίου πήραμε, λάβαμε πολλές ενδιαφέρουσες ε, ιδέες για μελλοντικού ελέγχους. Τώρα ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα εργασιών μας για το 2016 ως πρόγραμμα και έχουμε ήδη θεσπίσει τις προτεραιότητες σε έναν κατάλογο προτεραιοτήτων, task list. Τις επόμενες εβδομάδες θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα λοιπόν όπως σας ανέφερα για το 2016 και θα διαβιβαστεί στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου για την παρουσίαση τέλος αυτών των εκθέσεων, ιδίως των ειδικών εκθέσεων, special reports. Όπως γνωρίζετε πάντα παρουσιάζουμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού αυτές τις ειδικέ εκθέσεις. Ως τμήμα όμως της στρατηγικής μας να βελτιώσουμε τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, αρχίσαμε παρουσιάζοντας αναπερίπτωση αυτές τις ε, ειδικέ εκθέσεις στις ε, εξειδικευμένες κοινοβουλευτικές επιτροπές διευρύνοντας ε, το εύρος είναι πάρα πολύ σημαντικό ως στοιχείο βελτίωσης. Όμως το κύριο όφελος πρέπει να προέρχεται από το γεγονός ότι αυτή η εξειδικευμένη επιτροπή θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ευρήματα και τις συστάσεις μας όταν <clears throat> θα ε, γίνεται αποδέκτης νέων νομοθετικών προτάσεων και της εφαρμογής τους. Επιτέλους, η εξωτερική έλεγχη εξωτερικών ελεγκτών πρέπει να χρησιμοποιούνται πλέον στο πλήρες εύρος τους και τα σχόλια και αντιδράσεις του Ευρωκοινοβουλίου και στην ετήσια έκθεσή μας αλλά και στις ε, ειδικέ εκθέσεις και μέσω των ε, ψηφισμάτων. Μια και άλλαξαν οι καιροί πρέπει να εξετάζουμε πολύ καλύτερα πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα κονδύλια και έχει μίζωνα ρόλο να διαδραματίσει το Ευρωκοινοβούλιο σε αυτές τις διεργασίες. Ευελπιστώ ότι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει αυτού του είδους τις ειδικέ έκτακτες εκθέσεις στις δημοσιονομικές διαδικασίες αξιότιμα μέλη. Έχουμε δεσμευθεί να παράσχουμε αποτελεσματικά και φιλικά προς το χρήστη αποτελέσματα και στοιχεία. Χρειαζόμαστε τις δικές σας αντιδράσεις και παρατηρήσεις εφόλων αυτών των τριών πτυχών για τα όσα προτείνονται, πότε να υποβάλλονται αυτές οι προτάσεις και πώς να, να μπορούν να διαβιβαστούν και να αντιμετωπιστούν με το βέλτιστο τρόπο. Προσβλέπουμε σε αυτό το διάλογο μαζί σας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και εφεξής στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω ευχαριστώντας σας Πρόεδρε, εσάς την κοινοβουλευτική σας επιτροπή για αυτή την ευκαιρία αυτών των επαφών. Προσβλέπω σε οποιασδήποτε παρατηρήσεις ή οτιδήποτε έχετε να μας αναφέρετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σε τι να επικεντρωθούμε πότε να παράσχονται τα αποτελέσματα και το τρίτο μπορείτε να το επαναλάβετε άλλη μια φορά παρακαλώ αν θέλετε το τρίτο στοιχείο πώς να έχουμε την καλύτερη επικοινωνία σε αυτές τις επαφές μαζί σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Μπούζεκ Good. Ε, dear colleagues. Πολύ καλά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Κυρία, κυρία Ρίκουνεν, έχετε τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό το ερώτημα, το πώ ε, πρέπει να γίνεται αυτή η επικοινωνία. Και μια καλή αρχή για αυτή την επικοινωνία είναι ότι ήρθατε από το ελεγκτικό συνέδριο για να μα μιλήσετε. Είναι σημαντικό ε, να υπάρξει μια αλληλεπίδραση και εσείς να μας πείτε αυτό που θέλετε και εμείς αν μπορούμε να δώσουμε τη γνώμη μας. Καλό θα ήταν να μας εξηγήσετε περαιτέρω τα σχέδια που έχετε για το πρόγραμμα εργασιών 2016. Πού θα επικεντρωθείτε. Έχετε κάποιους ε, τομείς ε, που άπτονται με το πεδίο δραστηριοτήτων της Επιτροπής μας, ας πούμε, ενέργειας, έρευνας ή ε, βιομηχανίας. Και θα μας ενδιέφερε να μας πείτε δύο πράγματα παραπάνω για τα προβλήματα που εντοπίζετε και τους ε, λόγους, τις αιτίε που κρύβονται πίσω από αυτά τα προβλήματα. Είναι οι ασαφείς κανόνες, είναι πρόβλημα της νομοθεσίας. Ποιες είναι οι αιτίε ε, πίσω από τα προβλήματα που εντοπίζετε. Υπάρχουν διαφορές ε, μεταξύ κρατών μελών και έχετε εντοπίσει πιο συγκεκριμένου τομεί στους οποίους και εμεί θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπορέδη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο λόγια μόνο για να εκφράσω την εκτίμησή μου σε αυτό το όργανο, διότι θεωρούμε ότι είναι ένα όργανο που προσφέρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η καταπολέμηση της πατάλης των δημοσίων πόρων, η διαφάνεια, είναι ένα θέμα που αφορά το πολιτικό μας DNA. Είναι ουσιαστική σημασία λοιπόν να ενισχυθεί περαιτέρω η ανεξαρτησία του θεσμικού οργάνου τώρα πιο συγκεκριμένα ακόμα και αν φτάσαμε στο Κοινοβούλιο προενός έτους, ε, εκτιμήσαμε ιδιαίτερα κάποιες πρωτοβουλίε που αναλάβατε προσφάτως, να αναφέρω μόνο τρεις. Συνεχής έλεγχος που ποτέ δεν έπαψε για τις ασάφειες της Κομισιόν Μπαρόζο 2 για το εξαίρεση του προπολογισμού, ε, ο έλεγχος ορισμένων ευρωπαϊκών οργανισμών που εντοπίσατε διάφορα διαφορετικά προβλήματα μεταξύ των οποίων σύγκρουση συμφερόντων και προτείνατε ε, λύσεις ε, και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας ε, στα ό,τι αφορά τα ταμεία ε, συνοχής. Γνωρίζετε ότι το Ευρωκοινοβούλιο επιθυμεί αυτή η έλεγχη να ενταθούν και δίχως καμία προϋπόθεση. Αυτό που στο συμφέρον της Ένωσης και των πολιτών. Τέλος, βλέποντας τον σημαντικό ρόλο στην εθνική της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε βέβαιοι ότι το, οι, ε, σας οι δικοί σας ε, προσπάθειες θα είναι απαραίτητες για τον έλεγχο των οργάνων και των οικονομικών της Ένωσης. Θα στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία που θα λάβει προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. <clears throat> Uh, thank you, Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Θα ήθελα όχι να σας υπενθυμίσω, αλλά να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Πίτελα πολύ ορθά ανέφερε ότι η τακτική συνάντηση που γίνεται συνήθως είναι μια συνάντηση με την ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, τη CCC, στην οποία και παρέστη κατόπιν πρόσκλησής μου πριν από μερικούς μήνες. Όμως, αυτό ήταν το το καινούριο μάλλον, ε, είναι να έρχεται σε επαφή το ελεγκτικό συνέδριο με επιμέρους επιτροπές που έχουν ιδιαίτερη σημασία από πλευράς ε, ελέγχων και επιδόσεων του ελεγκτικού συνεδρίου. Γι' αυτό και τον ε, προσκάλεσα, γιατί θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα θετικό προηγούμενο. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος θέλει να λάβει τον λόγο. γιατί έχω και εγώ ορισμένα ερωτήματα. Προς τον κύριο Ήταλα. Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως τα πιο συχνά σφάλματα στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτά που εσείς θεωρείτε χαρακτηριστικά και συνήθη. Γιατί είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε. άλλο ζήτημα, όπως ο Horizon 2020 και το πρόγραμμα COSME. Η Επιτροπή ξεκίνησε τις προκατακτικές εργασίες για την ενδιάμεση αναθεώρηση και θα θέλαμε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι κι εμείς και για την ενδιάμεση αναθεώρηση, ιδίω ε, του ορίζοντα 2020, γιατί είναι δική μας ε, αρμοδιότητα να συμβάλλουμε και στην έκθεση της ε, Κομισιόν. Αν μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε σε αυτό το εγχείρημα. Τώρα όμως, όχι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τη Επιτροπής, αυτό θα ήταν πολύ καλό για μα. Αυτά. Okay. Any other requests for, for floor? Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τα ερωτήματά σας. Θα ξεκινήσω από τα δικά σας πρώτα. για το κόσμο και το πρόγραμμα Horizon 2020. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι όλες οι επιτροπές μπορούν πάντα να ζητούν τη γνωμοδότησή μας. Όπως ισχύει και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπως και τώρα που έχουμε αυτή την ενδιάμεσα αναθεώρηση αυτών των προγραμμάτων. Εγώ σας παροτρύνω, αν θεωρείτε ότι αυτό θα σας βοηθήσει, ε, μπορείτε βεβαίω να το κάνετε, να μας ζητήσετε. Είναι σημαντικό λοιπόν αν εσεί έχετε αυτή την άποψη. Αλλιώ δεν έχει νόημα εμεί να κάνουμε κάτι χωρίς να ξέρουμε αν σα ενδιαφέρει ή όχι. Και αν θα το την υπόψη ή όχι. Για αυτά τα προγράμματα όπως ο Ρίζον 2020 και το κόσμο δεν έχουμε ασκήσει έλεγχος προς την ε, υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων, γιατί βρίσκονται σε πρώιμα στάδια εφαρμογής τους. Δεν έχουμε και πολλά να ελέγξουμε δηλαδή ακόμα. Όμω, εκφωνήσαμε γνωμοδότηση τον Οκτώβριο του 2012 κατόπιν ετοίματο του Συμβουλίου για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα προγράμματα του ορίζοντα 2020. Βεβαίως πρέπει να επικαιροποιηθούν όλα αυτά. Στην ετήσια έκθεση για το 2014, που θα ε, δημοσιευθεί εδώ στο Κοινοβούλιο στις 10 Νοεμβρίου, θα δούμε πώς ε, οι στόχοι ε, των, του 2020 αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα συνοχής των κρατών μελών. Και θα εντοπίσουμε και κάποιους ε, κινδύνους και προκλήσεις ό,τι αφορά την εφαρμογή του ορίζοντα 2020. Αυτά για τον επόμενο μήνα. Μετά υπάρχει ένα σχεδιασμός, αλλά μόνο σχεδιασμός προς το παρόν, η ετήσια έκθεση για το 2015, η οποία βεβαίως θα δημοσιευθεί το 2016, να εξετάσει πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαχειρίζεται την ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 ιδίως ό,τι αφορά ε, τον ορίζοντα 2020, σε ό,τι αφορά τους στόχους και τα αποτελέσματα. Μετά, με ρωτήσατε τι είδους ε, σφάλματα εντοπίζουμε. Είναι πολλές διαφορετικές κατηγορίες. Πρώτον, συνήθως, αυτό αφορά τις αιτήσει εκθέσεις. Όμως πρόκειται για επιλέξιμες δαπάνες στις αιτήσει δαπανών. Για παράδειγμα, ΦΠΑ που θα μπορούσε να είχε επιστραφεί. Αυτό είναι σύνηθες. Μετά, για τα επιλέξιμα προγράμματα και τους δικαιούχους. Όπως είναι η καινοτόμο στήριξη για μη καινοτόμα προγράμματα. Επίση, πρόκειται για στήριξη που δίνεται σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ το κριτήριο είναι να δίνεται σε μικρές. Και βεβαίω υπάρχουν σφάλματα που σχετίζονται με τις δημόσιες προμήθειες. Και εδώ έχουμε πολλά παραδείγματα. Η αλλαγή του εύρου ε, τη σύμβαση εκ των υστέρων. Όμω ε, στι εξειδικευμένε μα εκθέσει εξετάζουμε κατά πόσο το πρόγραμμα επιφέρει προστιθέμενη αξία για την Ένωση και κατά πόσο τα χρήματα αυτά δαπανώνται αποτελεσματικά. Τώρα αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο και στη CCC και μετά να δούμε ποια είναι τα ζητήματα και τα θέματα στα οποία μπορούμε να ασκήσουμε έλεγχο. Βεβαίως δεν έχουμε και τόσους πόρους για να καλύψουμε όλα τα σημεία που ενδεχομένως να επιθυμούσαμε, όμως πρέπει να επιλέξουμε κάποια στοιχεία στα οποία θα επικεντρωθούμε αξιοποιώντας και τα διεθνή πρότυπα. Ας πούμε, τώρα θέλουμε να πιάσουμε το προσφυγικό. Και εκεί πρέπει να εξετάσουμε κάποια ζητήματα και να τα διαβιβάσουμε και στο Κοινοβούλιο. Όμω αυτή η συζήτηση για το πώ θα συνδράμουμε το Κοινοβούλιο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βεβαίω οι επιτροπέ μα ε, συνεχίζουν τη συνεργασία του, όμω ε, πολύ συχνά οι καλέ πληροφορίε και συστάσει για τι επιτροπέ εμπειρογνωμόνων είναι κάτι πολύ θετικό. Για να μπορούν να γίνουν και ιδιαίτερε συζητήσει εδώ στι εξειδικευμένε επιτροπέ. Ερωτήσετε, ποιες είναι οι επόμενες εκθέσεις στα τέλη της χρονιάς και για την επόμενη χρονιά. Μία τα αναφέρατε κι εσείς, βελτίωση της ασφάλειας, της ενεργειακής ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης της ε, ενιαίας αγοράς ενέργειας. Βεβαίως αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να το εξετάσουμε. Και τον Ιανουάριο του 2016 κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ένα κατάλληλο όχημα για την καινοτομία στην Ευρώπη. ή μάλλον το EIT για την καινοτομία και την τεχνολογία. Και μετά τον Ιούνιο του 2016 έχετε μια έκθεση που μας ενδιαφέρει και μετά δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει εσάς πολιτική για τα βιοκαύσιμα της Ένωσης. Βεβαίως είναι για την ένβη κυρίως αυτό το ζήτημα, αλλά ίσως και σας να σας ενδιαφέρει. αλλά και τα εμπορεύματα που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς, αλλά αυτό και ε, βεβαίω ε, αφορά την τραν. Όμως μπορείτε να εξετάσετε κάποια στοιχεία αυτών των ειδικών εκθέσεων. Αυτό απορρέει και τη δική μου εμπειρία. Όταν ήμουν ε, μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό είχα διαπιστώσει. Πρέπει να έχει κάποιο δύο, το πολύ τρει ειδικέ εκθέσει εκθέσεις κάθε χρόνο. Ευχαριστώ. Μία επιπροσθέτη ερώτηση από πλευρά μου. Υπό ποιες συνθήκες πρέπει ή μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σφάλματα, γιατί αναφερθήκατε πολλές φορές στον όρο σφάλμα, error. Μπορούμε, πρέπει να τα εξετάζουμε και να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα σφάλματα ως απάτη. Υπό ποιε συνθήκε. Και μετά ο κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω τις εξή ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν είναι ζητήματα δικής αρμοδιότητας, αλλά έτσι μου φαίνεται. Όταν ε, κάνετε αυτούς τους επιτόπιους ελέγχους, μιλήσατε και ε, για την βούληση των μικρών επιχειρήσεων. Πολύ συχνά από αυτές τις μικρές επιχειρήσεις μαθαίνουμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο σύνθετη είναι η διαδικασία να έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, ξεπερνά ακόμα και τις ανθρώπινες δυνάμεις κάποιες φορές. Πρέπει κάποιος ε, ε, να προσλάβει έναν μηχανικό, έναν τεχνικό υψηλού επίπεδου και υψηλών δεξιοτήτων για να αποκριτογραφήσει αυτά τα ζητήματα και αυτές τις απαιτήσει. Επίσης, η στιγμή που γίνεται, από τη στιγμή που γίνεται η αίτηση μέχρι την τελική εκταμείευση των κονδυλίων είναι πολύ μεγάλη χρονική περίοδος. Και πολύ συχνά αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικέ δυσκολίε αυτέ οι επιχειρήσει, ακόμα και κλείνουν τι πόρτε, γιατί καθυστερεί πάρα πολύ η εκταμίευση. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει απλούστευση εδώ, γιατί είναι κάτι το οποίο αναφέρουμε πολύ συχνά, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για το τέρα του Λόχνε. Όλοι γι' αυτό μιλάμε, αλλά κανεί δεν το βλέπει. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει δέσο επιμέλεια και γι' αυτό. Και Αυτός είναι και ο κύριο ε, ρόλος τη Ευρώπη εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα. Βεβαίω, εσεί λαμβάνετε τι αποφάσει. Εμεί εξετάζουμε αυτά τα ζητήματα και κάνουμε ειδικέ εκθέσει για να σας βοηθήσουμε. Κάποιες αφορούν τις μικροψηφίες επιχειρήσεις σας τα ανέφερα και προηγουμένως. Όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, ήδη τη δημοσιεύσαμε πριν από μερικούς μήνες. Και αφορούσε ακριβώς αυτό, πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να εξοπλίσουν αυτά τα ειδικά κονδύλια για να βελτιώσουν ε, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και άλλες εκθέσεις έχουμε δημοσιεύσει για τις μικρές επιχειρήσεις. Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τους μικροεπιχειρηματίες. Η γραμματεία μας ε, κάνει και το σχεδιασμό και μπορείτε να δείτε όλο τον κατάλογο μετά. μπορεί μετά ο εισηγητής που έχει αναλάβει αυτό το θέμα ε, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Μετά, για το θέμα της απάτης. Τα σφάλματα δεν συνιστούν απάτη. Πέρυσι, στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών μας, ελέγξαμε 1.200 ε, συναλλαγές με 14 περιπτώσεις που ενδεχομένω να αποτελούσαν απάτη. Και πάντα στέλνουμε αυτές τις περιπτώσεις στον Όλαφ και εκείνοι ανεξάρτητα αποφασίζουν τι θα κάνουν. Όμως πρέπει να κάνουμε μια διάκριση με τις περιπτώσεις απάτης. Βεβαίως, είναι προφανές. Τρία ερωτήματα από πλευρά σα. Σε τι να επικεντρωθούμε, απαντήσατε εν μέρη. Ποια είναι τα αποτελέσματα. το ΚΟΚΟΒΟΥ, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Κοκομπού ΚΟΚΟΒΟΥ ή ΚΟΜΤ είναι η προτεραιότητα και βεβαίως και η Επιτροπή μας και η Γραμματεία μας θέλει να ενημερώνεται και αν υπάρχει δυνατότητα θα σας προσκαλέσουμε και για περαιτέρω συζητήσεις εν ευθέτω χρόνο. Και για το τρίτο ζήτημα, πώς μπορεί να βελτιωθεί η επικοινωνία μας. Να κάνουμε άλλη μια συνάντηση και να υπάρξει επαφή με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι Επιτροπή αρμόδια για αυτά τα ζητήματα. Αν όμως χρειαστεί, θα υπάρξει και περαιτέρω συνάντηση. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις εξηγήσεις σας και προβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία με το Ελληνικό Συνέδριο. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκλώσαμε το πρώτο σημείο. Το δεύτερο είναι απαιτεί ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα περιμένουμε μέχρι τις 10.00, δηλαδή 20 λεπτά. Ο κύριος Έλμερ έχει το λόγο. Διαδικαστικό, από ό,τι κατάλαβα. Θέλω να αναφερθώ στην πρόταση των συντονιστών για την ε, ζήτημα της ανάθεσης των εξαίσεων Υπήρξε, ένα, υπήρξε που απασχόλησε πολλά, μέρη, πολλά μέλη, ειδικά από τη δική μας ομάδα. Θα ήθελα να στηρίξω τα όσα δήλωσε ο κύριος Τεμπεράνο ε, ευλόγω στις ε, περασμένες εβδομάδες. Ανησυχούμε, διότι το προηγούμενο σύστημα νομίζουμε ότι παρέχει σταθερότητα και ασφάλεια. Το νέο σύστημα θα το, δεν θα το πετύχει αυτό και θεωρούμε το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να ε, προκαλέσει διακρίσεις εις βάρος των ε, μικρών πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι αυτό παραβιάζει την ε, δημοκρατία στον οίκο μας. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να στηρίξουν τροπολογίες που έχει υποβάλει ο κ. Τεμπράνο και άλλοι, συμπεριλαμβάνουμε και την κυρία Μπάρβαρα Κέμπελ, όταν θα φτάσουμε στην ψήφιση αυτής της πρότασης. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Οι συντονιστές μας ε, αναφίβολα θα τα λάβουν υπόψη τα, αυτά που μόλις δηλώσατε. Θα ξεκινήσει λοιπόν η συνεδρίασή μας στις 30 αυτή των συντονιστών. Αυτά. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν για τις ψηφοφορίες. Uh, dear ladies and gentlemen, we've got a lot of uh, voting in front. και κύριοι, μας περιμένουν πολλές ψηφοφορίες. Δεν νομίζω πως θα τα καταφέρουμε να τελειώσουμε μέχρι τις 11. Λυπάμαι. Γι' αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ αμέσως. Θα μας χρειαστεί λίγο παραπάνω από μία ώρα. Πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. Ξεκινάμε λοιπόν με μια, έναν έλεγχο των ψηφοφορίας. Πάρτε όλε τις κάρτες σας παρακαλώ. Τοποθετήστε, τοποθετήστε στο, στο μηχανάκι. Και η ερώτηση έχει ως εξής. Σας αρέσει η συνεδρία της Επιτροπής μας σήμερα στο ημικύκλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Has anybody voted? Ψήφισαν άπαντες. Πέρα της εφορίας. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Και τώρα περνάμε στην πρώτη έκθεση. Μετά από τον έλεγχο που κάναμε μέσω του τεστ και ας ακούσουμε τώρα μερικά λόγια για τις χθεσινές ακροάσεις. Ε, ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, είχα την ε, ευχαρίστηση να σας αναπληρώσω χθες στη συνεδριάση μας. Σε αυτό την ακροάση υπήρξαν τρεις ε, καθηγητές από την Ευρώπη υπήρξε ένα συνδικαλιστή που ταξίδεψε από μακριά αλλά δεν ε, παρευρεθήκαν πολλοί συνάδελφοι αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα πρόκειται για ένα θέμα έλλειψης ευγένειας αγένειας θα μπορούσα να πω δεν υπήρξε κανείς ε, παρόν από, αυτούς, από την ομάδα ε, η οποία είχε προτείνει τη διεξαγωγή αυτής της ακρόασης. Αυτό είναι το σημείο που θέλω να θέσω. Uh, Uh, Ο αντιπρόεδρος μας λοιπόν έχει απόλυτο δίκαιο. Διότι αν προτείνουμε διεξαγωγή ακρόασης και προσκαλέσουμε σημαντικούς ομιλητές να έρθουν εδώ στο Κοινοβούλιο, είναι υποχρέωσή μας να παρευρεθούμε στην ακρόαση. Συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στην πρώτη έκθεση προς ψήφιση για την διαλειτουργικότητα θέμα των επιχειρήσεων και των πολιτών ίσα δύο διαλειτουργικότητα για τον εξορονισμό του δημόσιου τομέα. Συγητής Κάρλος Ζωρίνιο μία ονομαστική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Μόνο μία ψηφοφορία. Άρχιτη ψηφοφορία. Has, has everybody voted? Ψήφισαν άπαντες. Πέρα ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Ευχαριστώ τον εισηγητή. συζητήθηκε το θέμα ανάμεσα σε τρία θεσμικά όργανα και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση στο ίντερνετ οικουμενική υπηρεσία η συγητής μας η κυρία Πιλάρ Δεκαστήγιο υπήρξε μια έντονη συζήτηση και τώρα υπάρχουν συστάσεις ε, για δεύτερη ανάγνωση. Άρχεται ψηφοφορία. Has everybody voted? Ψηφίσατε πέρα της ψηφοφορίας. Σαφές ε, το αποτέλεσμα και εδώ. Σε χαρτίρια προς την εισηγητρία. Επόμενο θέμα τελική ψηφοφορία σχετικά με την ανάπτυξη μιας βιομηχανίας αηφόρου, ε, μιας αηφόρας βιομηχανίας για τα μέταλλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμβαστική πρόληψη 50, 15 συγγνώμη, θα μπορούσαμε να έχουμε μια ονομαστική ψηφοφορία. Εντάξει. Θα το έχω υπόψη μου. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ κατά εποχές δεκτή τροπολογία 4 και 12 ταυτόσιμες ομού υπέρ κατά εποχές δεκτές τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 και 14 ομού υπέρ, υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ <clears throat> κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για την 23. Πέρα ψηφορίας έγινε δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικός επί 24 Πέρα τις 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελεκτρονικά ψηφίζουμε την 27. Πέρα της <clears throat> Έγινε δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε ψηφίσουμε ηλεκτρονικός την 37 Οι S&D έχουν ένα πλέον ε, μέλος ψηφίσει ψηφίζει, πέρασε οι Δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικός άρχιτη ψηφοφορία, πέρα ψηφοφορίας. Δεκτή. 69 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε 69. ψηφίσμα. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 73 υπέρ κατά αποχές έλεγχος πέρα ψηφορίας ένας από το ΕΛΚ παραπάνω ψηφίζει πέρα ψηφορίας απορρίπτεται 74 υπέρ κατά ηλεκτρονικά θα ελέγξουμε 74 Υπέρ ψηφορίας δεκτή 75 υπέρ κατά αποχές δεκτή 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81, 82, 83, 85 και 82 υπέρ κατά αποχές δεκτής. Α, υπάρχει προφορική τροπολογία των πρασίνων. Αντικαθιστά αντικαταστήσει τον ε, Eurospace Industry ε, με το Transport Industry. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ. 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Συμβεστική. Υπέρ. 86 απορρίφθηκε. Α, ας επαληθεύσουμε. Επαληθεύουμε την 86. απορρίπτεται. Άξιζε τον κόπο να ελέγξουμε, δεν υπήρχε πάλι φορά. Συμβαστική τροπολογία, υπέρ κατά αποχές, ε, επαλήθευση, ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρα ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Εβδομήντα είναι υπέρ. Κατά εποχές 9 ψηφίζουμε ηλεκτρονικός 79 άρχιτη ψηφορία πέρασε δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές δεκτή 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές ας επαληθέψουμε 91 άρχιτη ψηφοφορία πέρας δεκτή 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 94 υπέρ κατά αποχές ας επαληθεύσουμε 94 άρχιτη την ψηφοφορία πέρασε απορρίφθηκε 125 υπέρ κατά αποχές Εκτή. 95 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ηλεκτρονικά 95 πέρα ψηφοφορίας δεκτή συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Ναι, ας επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 10. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 10. Πέρασε ο Απορρίφθηκε. Άξιζε τον κόπο να ελέξουμε. Ευχαριστώ για την παρατήρηση. Τροπολογία 88. Υπέρ.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 I 92 is adopted. Okay. Λοιπόν, εντάξει. Τροπολογία 88. Δεν την ψηφίσουμε. πίπτη 96 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές δεκτή 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή 110 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 110 άρχεται Electronic check. One... Ηλεκτρονικός έλεγχος, τροπολογία 110. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Απορρίφθηκε λοιπόν. Συμβιβασμός 11 υπέρ κατά αποχές δεκτός. Τροπολογία 106 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το συμβασμός 12 υπέρ κατά αποχές δεκτός 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβασμός 13 υπέρ κατά αποχές δεκτός δεν είναι εύκολο. Πρέπει να το ελέγξουμε. Δεν ήταν σαφές. Συμβασμός 13. Ψηφίζουμε το συμβασμό 13 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτός. <clears throat> Τροπολογία 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 138 υπέρ. Κατά θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 138. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 14 υπέρ κατά αποχές. Δεκτός. Τροπολογία 146 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. Τώρα έχουμε το συμβασμό 15 του ΕΛΚ που ζήτησε όμως ονομαστική ψηφοφορία. <clears throat> Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι σας πέρας ψηφοφορίας. Δεκτός ο συμβιβασμός 15. Στη συνέχεια τροπολογία 156 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 16 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτός. Τροπολογία 159 υπέρ, 159 υπέρ κατά αποχές δεκτός συμβασμός 17 υπέρ κατά αποχές δεκτός 165 166 ταυτόσημες ψηφίζουμε ομού υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε ψηφίζουμε την 156 και 166 165 και 166 ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας δεκτές. Συμβασμός 18 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τον συμβασμό 18. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε 170 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 170 άρχεται πέρας ψηφοφορίας δεκτή 171 υπέρ καταπίπτει λέτε καταπίπτει η 171 καταπίπτει εντάξει 174 και αυτή 175 υπέρ κατά Πρόεδρε, μπορείτε να εξηγήσετε γιατί 171 καταπίπτει. Η 171 καταπίπτει διότι η 170 είχε εγκριθεί, εγκρίθηκε η 170 και γι' αυτό αν η εγκριθεί η 170 η 171 καταπίπτει. 173 καταπίπτει, 174 καταπίπτει, καταπίπτουν αυτές. Ψηφίζουμε την 175 και μετά την 172. Τώρα η 175 λοιπόν, υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε, ψηφίζουμε την 175 ηλεκτρονικά, άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 172. 172 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 169 υπέρ. 169. Λοιπόν, 169 υπέρ, κατά, απόχες, απορρίπτεται. 176 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 176 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Θεέ μου. 177 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 177. Ηλεκτρονικός έλεγχος στην 177. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Συμβασμός 19 υπέρ κατά αποχές δεκτός 181 υπέρ κατά αποχές δεκτή 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή 190, 91, 92, 93 από κοινού όλες μαζί υπέρ αυτών κατά Απορρίπτονται. Θα ελέγξουμε λοιπόν. Ελέγχουμε αυτές τις τροπολογίες και τις ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται. Τέσσερις τροπολογίες λοιπόν. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτές. Μάλιστα. Συμβασμός 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. 199 υπέρ. Κατά απόχες. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 199 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 21 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτός. Τροπολογία 217 υπέρ. Κατά. Απόχες δεκτή αλλά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά 217 πέρας ψηφοφορίας τώρα δεκτή Θεέ μου 218 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε 218 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 219 υπέρ κατά απόχες απορρίφθηκε 220 υπέρ κατά απόχες δεκτή 222 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 222 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας αποτέλεσμα δεκτή Συμβασμός 22 υπέρ κατά αποχές δεκτό. Συμβασμός 23 υπέρ κατά αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε τον συμβασμό 23 ηλεκτρονικά άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε ο συμβασμός 23. 229 και 230 από κοινού. Υπέρ αυτών. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε και τις δύο. 229-230 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτές. 225 εντάξει και η 225 πολύ καλά 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 233 ηλεκτρονικά άρχεται Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτός. 244 τροπολογία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει λέγεται στον πρόεδρο. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Επειδή έχουμε το συμβιβασμό 24 δεκτό στο δεύτερο τμήμα τώρα αυτό στην 244 καταπίπτει 241-242 ομού είναι ταυτόσιμες υπέρ αυτών κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε αυτές τις δύο τροπολογίες 241-242 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας δεκτές συμβασμός 25 υπέρ κατά αποχές δεκτός. Συμβασμός 26 υπέρ, κατά αποχές δεκτός. 247 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 27 υπέρ, κατά αποχές δεκτός. 251 υπέρ, κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 251 ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Η ισοψηφία απορρίπτεται. απορρίφθηκε. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 253 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 253. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 261 υπέρ κατά αποχές δεκτή 262 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 262 άρχεται πέρας ψηφοφορίας δεκτή συμβασμός 28 υπέρ κατά αποχές δεκτός τροπολογία 263 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 263 άρχεται ελέγχουμε ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε συμβασμός 29 υπέρ κατά αποχές Νομίζω απορρίφθηκε, αλλά θα ελέγξουμε. Την ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τον συμβιβασμό 29 δηλαδή. 29. Πέρας ψηφοφορίας και αποτέλεσμα δεκτός. Δεκτός. Και τελική ψηφοφορία τώρα που φυσικά θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας δεκτή. 47 υπέρ 11 εναντίον 3 αποχές. Συγχαρητήρια στον ε, εισηγητή μας κύριο Εντουάρντ Μαρτάν. Πολύ καλά. Και τώρα έχουμε την έκθεση του κυρίου Λεβαντόφσκι. Κεφαλαιακή αγορά, Ένωση Κεφαλαιακών Αγορών. Πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, ενωσιακό πλαίσιο για τις διατάξεις ε, χρηματοοικονομικές διατάξεις. Απολογισμός και προκλήσεις ε, των ε, ρυθμίσεων για τις υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Λοιπόν, πολύ καλά. Ξεκινάμε λοιπόν. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Τροπολογία 1. Ψηφίζουμε την τροπολογία 1. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Συμβασμός 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτός. Τροπολογία 7. Πρώτο τμήμα. Σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε το πρώτο τμήμα. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 7 πρώτο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτό το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Καταπίπτει αυτό. Επειδή ο συμβασμός 1 εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε 11 υπέρ κατά θα ελέγξουμε την 11 άρχεται πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές δεκτός τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές δεκτός. 29 υπέρ κατά αποχές δε, απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 31 άρχεται 31 πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε σαφέστατο το αποτέλεσμα 32 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να ελέγξουμε να σηκώνετε ξεκάθαρα τα χέρια σας 32 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας δεκτή παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας για να μπορούμε να δούμε πως ψηφίζετε 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ Καλά. Κατά. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 34. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτός. Προπολογία 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε την 48. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 49 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίφθηκε. 50 υπέρ. Κατά Θα, ψηφ, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά προς έλεγχο την 50. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή η 50. Να σηκώνετε καθαρά ξεκάθαρα τα χέρια σας. Ξέρω, έχετε κουραστεί. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. 51. Ηλεκτρονικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 52 υπέρ κατά Α, δεν μπορούμε να δούμε το αποτέλεσμα 52 ηλεκτρονικά άρχεται πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε 53 υπέρ κατά άποχες απορρίφθηκε 54 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές δεκτός 58 είχαμε έτοιμα της ε, ΓΚΟΕ της Ενωτικής Αριστεράς για ξεχωριστή ψήφιση μετά από έτοιμα λοιπόν της ΓΚΟΕ η 58 τροπολογία ψηφίζεται ξεχωριστά υπέρ αυτής κατά αποχές απορρίφθηκε Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. 63 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 64 υπέρ κατά απόχες δεκτή 66 υπέρ κατά απόχες δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 68 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 69 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 70 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 70 άρχεται ελέγχουμε ψηφίζοντας ηλεκτρονικά πέρας ψηφοφορίας δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ψηφίζουμε την 72 άρχεται πέρας ψηφοφορίας απορρίφθηκε και τώρα η τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία άρχεται Ψηφίσατε όλοι. Ένας από το ΕΛΚ παραπάνω, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Αποτέλεσμα. 50 υπέρ. 8 εναντίον. 6 αποχές. Συγχαρητήρια συνάδελφε Λεβαντόφσκι, Γιάννους Λεβαντόφσκι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στην τελευταία ψηφοφορία που έχουμε. Προφορική ερώτηση. Προφορική ερώτηση για την οικονομία με βάση τα δεδομένα της ε, κυρίας Μπάρμπαρα Κάπελ. τελική ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία για το προφορικό ερώτημα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με πέντε αποχές. Και 39 υπέρ. Τώρα, πρόταση ψηφίσματος για μια ευημερούσα οικονομία με βάση τα δεδομένα. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική τρία, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τέσσερα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πολύ περίπλοκη ψηφοφορία. Ιδίω για τους σοσιαλδημοκράτες. Ήμικο Β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήμικο Σ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί 42 πέρας απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 49 Πέρας. Α, συγγνώμη. Δεν έβλεπα τα χέρια σας. Λοιπόν. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σημαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική βεβαίω το 19. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 70 πέρας απορρίπτεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Την 156. Πέρας. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Σεβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 164 υπέρ. Α, 164 και 165 ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε και τις δύο λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 182. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 182. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2.37. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίβεται. Συμβαστική 28. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά τη συμβαστική 28. Για να σιγουρευτούμε.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 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, ναι, συγγνώμη. Πριν τη 39 πρέπει να ψηφίσουμε τη 2.28. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, συμβαστική 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 2.35. Πέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.41. Υπέρ κατά αποχές Ας ελέγξουμε τη 2.41 2.49 συγγνώμη Α, 2.41 διορθώνει ο πρόεδρος Πέρας Απορρίπτεται Συμβαστική 40 υπέρ Κατά Αποχές Εγκρίνεται 2.42 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ, 5 κατά, 9 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Κάπελ για την έκθεσή τη. Okay. <coughs> Now, dear colleagues, we've got uh, our coordinators. Λοιπόν, συνάδελφοι, έχουμε την συνεδρία των συντονιστών, αλλά για όλους σας είναι σημαντικό στις 3 το απόγευμα. Έχουμε κοινή συνεδρίαση δύο επιτροπών. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, να έχετε υπόψη σας λοιπόν ότι έχουμε κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΙΜΚΟ στις 3 το απόγευμα. Να είμαστε όλοι εδώ. Να έχουμε ισχυρότατη εκπροσώπηση της ε, Επιτροπής μας. Ε, δηλαδή 100% συμμετοχή. Ωραία, ευχαριστώ. Συνεδρία των συντονιστών τώρα.